θα προωθήσω τα ψηφίσματα που εθετήσαμε στα πρακτικά αυτά. Διακόπτεται η σύνοδος και λύεται η παρούσα συνεδρία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνήσεις.